με τις συνθήκες για διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας. Έκλεισε το μικρόφωνο του ομιλητή. Και θέλουμε να ε, βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας όλων των ε, εργαζομένων, κυρίως των νεοεισερχομένων και αυτών που δεν έχουν σταθερή θέση εργασίας. Επίσης ε, προσπαθεί να συμμορφωθεί, να προωθήσει μάλλον τη συμμόρφωση με τις συνθήκες εργασίας κατά την έννοια αυτή ε, θα πρέπει όσο γίνεται περισσότερο να κλείσουν ε, οποιαδήποτε κενά. Ε, θα πρέπει να υπάρχουν εγγυημένε ώρες εργασίας πληρωμένες και επομένως δεν είναι δυνατόν να επιτρέπουμε τη συνέχεια των λεγόμενων zero hour contract, των συμβολέων μηδενικών ωρών. Θα πρέπει η εργοδοσία να δίνει σωστές και συμπληρωματικές και ολοκληρωμένες μάλλον πληροφορίες για όλα τα στοιχεία γιατί διαφορετικά Υπάρχουν κίνδυνοι, διατρέχουν τον κίνδυνο να μην ε, καλύψουν τις υποχρεώσεις τους, αλλά να τις μετακυλήσουν σε ένα τρίτο ε, μέρος. Επίσης, οποτεδήποτε οι εργοδότες ε, πρέπει ε, να ε, πληροφορήσουν τον εργαζόμενο για, τις, για τα βασικά στοιχεία της εργασιακής σχέσης, οπωσδήποτε θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι στις πληροφορίες θα αναφέρονται τουλάχιστον οι βασικές πληροφορίες όσον αφορά την πάυση της συνεργασίας, καθώς επίσης και όλες οι ε, πράξεις οι οποίες σχετίζονται με την αποζημίωση σε περίπτωση πάυση της σχέση ή σε περίπτωση ή σε περίπτωση παραβίασης εργασιακών δικαιωμάτων. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης υποχρεώσεις ε, που θα αναφέρονται στην ε, υπέρβαση ωραρίου, καθώ επίσης ε, και οποιασδήποτε προσφυγέ ή παράπονο προκύψουν από τέτοιες υπερβάσεις. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι πάρα πολύ σημαντικά έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν πάντα την δυνατότητα να ασκήσουν τα δικαιώματά τους γνωρίζοντας και τα χρονικά περιθώρια, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι πολύ στενά. Επίσης, ε, οι πληροφορίες όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις και όλες τις λεπτομέρειες που ανέφερα προηγουμένως θα πρέπει ε, να εγχειρίζονται στον εργαζόμενο ε, ή αλλιώς θα πρέπει να μεταδίδονται με ηλεκτρονική μορφή αλλά με επιβεβαίωση παραλαβής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οπωσδήποτε σε γλώσσα που κατανοούν οι εργαζόμενοι. Οι ξένοι εργαζόμενοι επίσης θα πρέπει με σαφήνεια και ε, αμεσότητα να ε, πληροφορούνται για όλα τα στοιχεία αυτά. Επίσης, ε, για να αποφευχθεί ε, η κακή χρήση μιας ε, περίοδου δοκιμασίας, θα πρέπει οποτεδήποτε μια εργασιακή σχέση υπόκειται σε τέτοια δοκιμαστική περίοδο, αυτή η δοκιμαστική περίοδος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Επίσης, τα κράτη-μέλη που είναι υποχρεωμένα να βρουν ισορροπημένες λύσεις μεταξύ των δύο ε, μερών θα πρέπει να ε, αναφέρουν συγκεκριμένες δυνατότητες μη συμμόρ... συγγνώμη, συγκεκριμένες περιπτώσεις μη ε, συμμόρφωσης έτσι ώστε να μην υπάρξουν ας πούμε συγκρούσεις συμφερόντων. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι δυνατόν να επιτραπεί στους εργοδότες μόνο μερός να ορίζουν κάποιες περιπτώσεις ασυμβατότητας είναι ξεκάθαρο ότι τα πρότυπα τα οποία αναφέρονται ε, σε, αυτήν την, ε, σε αυτό το κείμενο ότι δεν μπορούν να υπόκεινται σε συλλογικές συμβάσεις. Επίσης ε, θα πρέπει να αρχίσουν να παράγουν άμεσα αποτέλεσμα. Επίσης, η, επίσης θα πρέπει να προβλέπονται ρητές νομικές διαδικασίες ή νομικά αποτέλεσμα αποτελέσματα ε, σε σχέση με τα δικαιώματα τα οποία αναφέρονται σε τούτη την πρόταση. Ε, οι εργοδότες θα πρέπει να παράσχουν ε, αρκετές και ικανοποιητικές πληροφορίες όσον αφορά ιδιαίτερο στην απόλυση γιατί διαφορετικά δεν θα έχει νομική ισχύ η απόλυση. Όλα τα απαραίτητα μέτρα θα πρέπει να ληφθούν έτσι ώστε οι προθεσμίες ε, για δυνατότητα ε, άσκησης προσφυγής ή αντίρρησης. Ε, οι προθεσμίες, λέω, δεν θα αρχίσουν να μετρούν παρά μόνο από τη στιγμή που θα έχει λάβει ρητή γνωστοποίηση για την απόλυση ο εργαζόμενος. Τέλος, ε, θα πρέπει ρητά να αναφερθεί ε, ότι η υλοποίηση ε, και η θέση εφαρμογή της οδηγίας του κανονισμού αυτού συγγνώμη, δεν θα αποτελέσει προηγούμενο για ανέρεση οποιονδήποτε στοιχείων αναφέρονται στη, στα γενικά επίπεδα προστασίας των δικαιωμάτων στα κράτη-μέλη και οπωσδήποτε κανένα επίπεδο προστασίας ε, δεν θα πρέπει βάσει του κειμένου αυτού να μειωθεί. Αντιθέτως ε, θα πρέπει οπωσδήποτε ε, ρυθμιστικά να βελτιωθεί η προστασία των εργαζομένων στα πλαίσια του πεδίου εφαρμογής του εν λόγω κειμένου λαμβάνοντας υπόψη και τα όσα αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Χάρτα. Επίσης, θα πρέπει να γίνει έργο ε, το ε, άρθρο της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που αναφέρει ότι ο κάθε ένας εργαζόμενος έχει δικαίωμα ε, για καλά αμοιβόμενη και αξιοπρεπή εργασία. Ευχαριστώ. Σχόλια παρακαλώ. Εγώ είμαι σκιώδης και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο κύριο Χρυσόγωνο για την ε, έκθεση, για την γνωμοδότησή του αυτή. Ε, και στις Βρυξέλλες ε, και στην Μάλτα έχω έρθει σε επαφή με πολλούς ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους και θα σε επαφή με εκπρόσωπους της εργοδοσίας αλλά και εργαζομένων ε, και μπορώ να σας μεταφέρω κάποια από τα στοιχεία τα οποία συζήτησα μαζί τους και τις σκέψεις που μου υπέβαλαν. Ας πούμε, όσον αφορά την ιδέα ότι θα πρέπει να υπάρχει γραπτή δήλωση και επομένως αφήνει εξ αρχής, πιστεύω ότι αυτό είναι θεμελιώδου σημασίας διότι συζητούμε τώρα ε, για ε, την δυνατότητα εξαίρεσης ε, για περίπτωση που ο εργαζόμενος εργάζεται λιγότερο από 8 ώρες την εβδομάδα. Αλλά αυτό στην ουσία είναι ένα μεγάλο κενό και πιστεύω ότι θα πρέπει η εξαίρεση να βασίζεται σε 8 ώρες εργασία ανά μήνα. Επίσης, ε, στην πρώτη περίπτωση δεν δίνεται η δυνατότητα ε, να ληφθούν υπόψη στοιχεία εποχικότητας ε, κλπ. Πιστεύω ότι εδώ έχουμε μια καλά ισορροπημένη πρόταση, γιατί βεβαίως θα πρέπει οπωσδήποτε να αποτρέψουμε οποιαδήποτε μορφή επισφαλούς εργασίας. Εάν ε, τώρα το γεγονός, ε, το θέμα μάλλον της, ε, του ενιαίου ορισμού του εργαζόμενου worker, έχουμε περιπτώσεις εργαζομένων που μετακινούνται από χώρα σε χώρα και επομένως καλό θα ήταν να υπάρχει ένας ευρωπαϊκός ορισμός. Όσον αφορά τις συμβάσεις, αυτές είναι όντως σημαντικές όχι μόνο για τον εργαζόμενο αλλά και για τον εργοδότη και ε, κατανοώ ότι ε, εδώ αναφερόμαστε ε, σε χάρτινο έγγραφο και όχι μονάχα γενικά έγγραφο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό έτσι ώστε ο εργαζόμενος να γνωρίζει ακριβώς τις συνθήκες και τις λεπτομέρειες που συνδέονται με την θέση εργασίας του εργαζόμενου ή της εργαζόμενης. Νομίζω ότι και σε αυτή την έννοια μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σωστά το θέμα με τη δημιουργία ενός template. Ένα άλλο θέμα, το οποίο το οποίο φαίνεται να απασχολεί όλους τους εμπλεκομένους, είναι το θέμα της υποχρεωτικής δωρεάν κατάρτισης. Είδαμε περιπτώσεις όπου ε, ε υπάρχουν άνθρωποι στη Μάλτα, ας πούμε, που προσπαθούσαν να ε, βρουν θέση εργασίας, να προσληφθούν τέλος πάντων ως προσωπικό καμπίνας αεροσκάφους ε, στην ε, Μάλτα και τους υποχρεώνουν να περνάνε από μια κατεύθυνση. Επίσης έχουμε τους Learning Support Educators που ε, τους ε, ζητούν να περάσουν από υποχρεωτική μεν εκπαίδευση, η οποία όμως δεν ε, καλύπτεται, θα πρέπει να την πληρώσουν από την τσέπη τους. Όλα αυτά είναι απαράδεκτα. Η κατάρτιση εφόσον είναι υποχρεωτική και από πλευράς του ιδιωτού εργοδότη, τότε οπωσδήποτε δεν θα πρέπει να επιβάλλει οποιοδήποτε κόστος, επιπλέον κόστος στον εργαζόμενο. Από την άλλη πλευρά, από πλευρά των ε, ε, εργοδοτών, θα πρέπει να υπάρχει κάποια εξασφάλιση ότι τα χρήματα, το κόστος ε, το οποίο αντιπροσωπεύει αυτή η κατάρτιση θα πρέπει με κάποιο τρόπο να επιστραφεί στον εργοδότη. Δηλαδή ότι αυτός ο εργαζόμενος θα πρέπει να παραμείνει για κάποιο διάστημα στον εργοδότη. Αυτά όσον αφορά τα διάφορα στοιχεία. Επίσης, ε, ε, οι έξι μήνες ε, νομίζω ότι είναι ένα καλό όριο, αλλά βεβαίως θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί και το ενδεχόμενο των τριών μηνών. Και από ό,τι καταλαβαίνω, η από ό,τι καταλαβαίνω, σε ορισμένες περιπτώσεις όπως και στην Μάλτα ε, εάν δεν υπάρχει καμία ε, ρητή αναφορά στο συμβόλαιο, ε, τότε αυτή η δοκιμαστική περίοδος θεωρείται ότι δεν υπάρχει ή ότι στο τέλος των έξι ή των τριών μηνών de facto ο εργαζόμενος ενσωματώνει στο προσωπικό της εταιρείας. Το ζήτημα είναι λοιπόν να δούμε ε, ε, ε, επίσης το θέμα της μερικής απασχόλησης και να υπάρχει σύγκρουση και να αναγνωρισμένη σύγκρουση συμφερόντων μονάχα σε ορισμένες πολύ συγκεκριμένες και ειδικές περιπτώσεις. Οι προκλήσεις είναι υψηλές εδώ, αλλά δεν είμαστε εμείς η Επιτροπή Απασχόλησης, συναδελφοί. Εμπάσπευτος, να κάνω μια συγκεκριμένη, θα έλεγα, παρατήρηση. Ο ορισμός του εργαζομένου δίδεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και πάρα πολύ αναλυτικά. Ε, δεν είναι το θέμα αν μας αρέσει ή όχι. Λοιπόν, αυτά. Δεν βλέπω κάποιον άλλον ο οποίος έχει ζητήσει το λόγο. Συνεπώς... στο συγκεκριμένο σημείο θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ως σκιώδης για το συγκεκριμένο θέμα θα ήθελα να κάνω κάποια πολύ σύντομα σχόλια. Πρώτον, θα ήθελα να πω ότι η πρωτοβουλία είναι πάρα πολύ θετική σε σχέση με την προβλεψιμότητα και τη διαφάνεια των συνθήκων εργασίας. Είναι κάτι το ιδιαίτερο θετικό. Ταυτόχρονα νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο την πρόταση αυτή, έτσι ώστε να είμαι θα ότι η οδηγία έχει όλα τα μέσα τα οποία απαιτούνται για να διασφαλίζει ακριβώς ένα πλαίσιο δίκαιο και διαφανές. Έχω την αίσθηση ότι ένα πιο ευέλικτο σύστημα εργασίας είναι θα έλεγα συμβατό με την κοινωνία την ψηφιακή στην οποία ζούμε και ένα τέτοιο ευέλικτο σύστημα θα μπορεί να αντιδράσει περαιτέρω αλλαγές και στο μέλλον. Νομίζω λοιπόν ότι ήδη στην αρχή της σύμβασης εργασίας και όχι για δύο μήνες όπως προεβλέπετο δεν είναι κακή η πρόταση αυτή βέβαια. Θα πρέπει επίσης να απαγορεύονται υπερβολικά μακρόχρονες δοκιμαστικοί περίοδοι κτλ. Νομίζω ότι οι προτάσεις ε, έτσι που γίνονται βελτιώνουν την αρχική πρόταση. Θα πρέπει λοιπόν οι προτάσεις μας να δίνουν ε, δίκαια πλεονεκτήματα και στον εργοδότη αλλά και στον εργαζόμενο. Η Επιτροπή θα ήθελε το λόγο. Όχι. Καλώς, ευχαριστώ. Στρέφομαι στον εισηγήτη. Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι 29 Ιουνίου. Λάβετε το υπόψη. Και κλείνουμε το θέμα αυτό, τη συζήτηση αυτή. Συνεχίζουμε με το 19. Ανταλλαγή απόψεων και εδώ. Την παρουσία των γνωμοδοτών για την προστασία αυτών οι οποίοι καταγγέλουν για λόγους ε, ε, παραβίασης του, ε, του ευρωπαϊκού δικαίου. Η κυρία Οζιέρ είναι η συγγήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που έχω μαζί σας αυτή την πρώτη συζήτηση για την πρόταση οδηγίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταρχάς θα πρέπει να είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι που ε, αυτή τη φορά εισακουστήκαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσης θα μπορέσουμε να ζητήσουμε, όπως και το κάναμε τον προηγούμενο Οκτώβριο, την προστασία των καταγγελόντων για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Οι προτάσεις τις οποίες έχουμε μπροστά μας περιλαμβάνει κάποιες από τις αρχικές μας προτάσεις της 24ης Οκτωβρίου του 2017. Παρακαλώ λίγη ησυχία. Επανέρχομαι στο περιεχόμενο της πρότασης. Καταρχάς για το πεδίο εφαρμογής. Εγώ εκφράζω την ικανοποίησή μου γιατί έχουμε ένα αρκετά φιλόδοξο πεδίο εφαρμογής στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάτι το οποίο παρέχει προστασία στους εργαζομένους αλλά και σε αυτούς που δεν έχουν άμεση σχέση με εργοδότες, δηλαδή συμβούλους, τέος εργαζομένους, ανεξάρτητους επαγγελματίες, σταζιέρ σχετικά με το πραγματικό τώρα, το υλικό πεδίο εφαρμογής. Κατανοούμε την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ανοίξει ορισμένους τομείς έτσι ώστε να καταλήξουμε στο λεγόμενο οριζόντιο μέσο. Όμως, αυτό θέτει κάποια θέματα σε σχέση με το πραγματικά οριζόντιο χαρακτήρα του μέσου και στην έλλειψη τομέων οι οποίοι θα μπορούσαν να καλυφθούν αλλά δεν καλύπτονται. Τίθενται ας πούμε κάποια θέματα σε σχέση με το κοινοτικό κεκτημένο για την προστασία των εργαζομένων. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί εξαιρείται από την οδηγία το συγκεκριμένο πεδίο. Μια άλλη ανησυχία είναι ότι το κείμενο αναφέρεται στις παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου. Ακούμε την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία θέλει να προστατεύσει από ε, αποκαλύψεις που θα φέρουν στην επιφάνεια κάποιες απάτες, αλλά ταυτόχρονα θέλει να καλύψει και κάποιες ε, ε, περιπτώσεις θα έλεγα οι οποίες παραποιούν την ισχύουσα κατάσταση στα ευρωπαϊκά όργανα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θέτει το πρόβλημα της παραβίασης του δημοσίου συμφέροντος. Κάθε πολίτης θα μπορούσε να βρεθεί σε μια κατάσταση να λειτουργήσει ως ε, μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος και ταυτόχρονα δεν θα είναι σε θέση να γνωρίζει το νομικό μέσο. Παρακαλώ τις κυρίες εκεί αριστερά να, να κάνουν ησυχία, ζητώ από τα μέλη της γραμματείας να κάνουν λίγη ησυχία. Ε, θα έλεγα λοιπόν ότι κάθε πολίτης δεν είναι σε θέση να γνωρίζει λεπτομερώς τον κοινοτικό νόμο και να γνωρίζει αν τα, αυτά για τα οποία κατηγορείται ε, εντάσσονται στη συγκεκριμένη νομοθεσία ή όχι, καλύπτονται από την νομοθεσία αυτή. Τώρα, εδώ ε, συγχαίρω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί θέλει και σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο των κοινοτικών οργανισμών ε, αυστηρά μέτρα και δημοσιοποίηση ε, για την ύπαρξη αυτών των προβλημάτων και αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Αυτό το οποίο όμως είναι προβληματικό, η λεγόμενη διάβλη καταγγελίας. Ε, επίσης ε, αυτό το οποίο δεν διευκρινίζεται είναι το πώς θα χρησιμοποιήσουν τους διάβλους αυτούς οι καταγγέλλοντες έτσι ώστε να υπάρξει μια σταδιακή χρήση τους, δηλαδή ένας εξωτερικός, εσωτερικός διάβλος πρώτα, ένας εξωτερικός κατά δεύτερον και από εκεί και πέρα κάτι το διαφορετικό. Προβλέπονται αποκλήσεις οι οποίες επιτρέπουν το να στρέφεται κανείς στους εσωτερικούς διάβλους ή στους δημόσιους διάβλους. Μιλάμε επίσης και για τους περιορισμούς του εσωτερικού διάβλου και αυτό για δύο λόγους. Καταρχάς, ο καταγγέλων είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να αποδείξει την ανάγκη να μην προσφύγει στον εσωτερικό διάβλο. Ο καταγγέλων υφίσταται υψηλότατες πιέσεις, πολλές φορές αμφισβητείται, καταγγέλλεται ε, το ηθικό της πράξης του κτλ. Συνεπώς λοιπόν εδώ στην ουσία κάνουμε ένα ακόμα βήμα για να του στερήσουμε το όφελος της προστασίας. Εμποδίζουμε λοιπόν τον μίσθωτο, ο οποίος γνωρίζει μια αυστηρή παραβίαση, να έρθει σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές. Ενώ στην περίπτωση μιας σοβαρής παραβίασης δεν χρειάζεται να υπάρξει εσωτερικός διάβλος, οι ρυθμιστικές υπηρεσίες είναι αυτές οι οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα μέσα τα οποία είναι διαθέσιμα και πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τους εξωτερικούς διάβλους και αυτή η σταδιακή χρήση των μέσων αποκλείει αν θέλετε το δικαίωμα στη γνώση ουσιαστικά ε, ορισμένων ε, προβλέψεων, διατάξεων που αφορούν την ύπαρξή μας ως πολίτες και ως προς αυτό ο καταγγέλων στην ουσία λειτουργεί ενημερωτικά για τους πολίτες. Τώρα σχετικά με την προστασία που είναι κάτι που ανήκει και στην προηγούμενη έκθεση του μηνός Οκτωβρίου. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπεριλαμβάνει τους δύο τύπους προστασίας, τη μισθολογική προστασία από τη μία και την προστασία επίσης δικαστικών διαδικασιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν πήρε θετικά τις απόψεις μας Επίσης το θέμα της απόδειξης, ε, της αναστροφής της ευθύνης ε, σε περίπτωση αντιμέτρων και επίσης η δυνατότητα βοήθειας νομικής ε, και διαδικαστικής τους καταγγέλλοντες. Εδώ θα ήθελα να πιέσουμε κάπως τα κράτη-μέλη για να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο τους καταγγέλλοντες. Νομίζω επίσης ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τις προβλέψεις της προστασίας της ταυτότητας του καταγγέλλοντος ε, έτσι ώστε να είναι επαρκής οι εγγυήσει για την προστασία αυτή. Και ένα τελευταίο σημείο. Εγώ δεν είμαι υπέρ της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κυρώσεις επιπροσώπων οι οποίοι θα ε, ξεκινούσαν διαδικασίες καταγγελίας με κακές προθέσεις. Έχουμε έτσι και αλλιώς εθνικούς νόμους που προβλέπουν την προστασία από συκοφαντική δυσφήμιση, απλή δυσφήμιση ε, κτλ. Ε, συνεπώς ε, δεν θα πρέπει να αποδυναμώσουμε εμείς τη θέση του καταγγέλλοντα, ο οποίος ε, ναι μεν δεν θα διώκεται για συκοφαντική δυσφήμιση, αλλά θα μπορεί να διωχθεί εσωτερικά. Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις σε σχέση με αυτά που είχαμε ζητήσει στο παρελθόν. Θα πρέπει οι αρχές δίωξης να νομιμοποιηθούν ακόμα περισσότερο διοικητικά ε, επί τη βάση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης το θέμα της ανωνυμίας δεν αντιμετωπίζεται. Ξέρουμε ότι η πλαισιούμενη δυνατότητα να υπάρχουν ανώνυμες καταγγελίες ε, μπορεί να μας βοηθήσουν να ανοιχνεύσουμε ορισμένες παραβιάσεις και αποσιωπούμε αυτούς που βοηθούν, στηρίζουν, συμβουλεύουν τους καταγγέλλοντες. Θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για αυτούς έτσι ώστε να μην υφίστανται αντίπεινα και αυτοί. Καλή η πρόταση γενικά. Χαίρομαι που η Επιτροπή δέχεται τις προτάσεις του Κοινοβουλίου. Μπορούμε να την βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο και αυτό θα κάνουμε με τους σκιώδεις εισηγητές Ελπίζω να ξεκινήσει η συζήτηση. Ευχαριστώ όλους για την προσοχή τους. Πρόεδρος, ευχαριστώ εσείς κύριε Τζιρόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα έχω να πω μόνο ότι προφανώς συμφωνώ την με την ανάλυση που έκανε η Βιρζινή. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έλαβε υπόψη το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Έρχομαι και λίγο πιο πίσω, δηλαδή ευχαριστώ και όλες τις πολιτικές ομάδες που έλαβαν υπόψη αυτό που είχαμε προτείνει. Θα θυμάσαι, Βιρζινία, από την αρχή το είχαμε προτείνει εμείς. Μετά από την ε, έγκριση της οδηγίας για το επαγγελματικό ε, απόρριτο. Χαίρομαι λοιπόν. Τώρα έχω να πω μονάχα ότι το ζήτημα της προστασίας της ανωνυμίας υπορισμένες συνθήκες εμένα μου φαίνεται αναγκαίο και το ίδιο θα χρειαστεί να συζητήσουμε και την μη ιεράρχηση των επιλογών των διάβλων που χρησιμοποιούνται ή που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καταγγελία ενός θέματος γενικού ενδιαφέροντος. Θα το ξανασυζητήσουμε, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και κάποιες... Ε, ε, μάλλον δεν υπάρχουν ορισμένες δυνατότητες. Και είναι σημαντικό το ότι δεν έχει ληφθεί υπόψη και το εμπρόθετο, το ζήτημα δηλαδή της ε, πρόθεσης. Και εκεί είναι σημαντικό πρέπει να ληφθεί υπόψη και από την Επιτροπή. Μάλιστα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Διδιέ. Ευχαριστώ πολύ την ε, Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια. Ω και ο εισηγητή του Λαϊκού Κόμματο, πιστεύω ότι πράγματι θα μπορέσουμε έτσι να προστατεύσουμε καλύτερα του καταγγέλλοντε. Ε, παρατηρώ εξάλλου ότι το σχέδιο οδηγία ε, εμπνέεται από το γαλλικό δίκαιο. Και γι' αυτό ίσω και τόσο πολλοί Γάλλοι όπω οι ε, εισηγήτρια και οι εισηγητέ είμαστε γαλλική επικότητα, είμαστε Γάλλοι. Και το Λαϊκό Κόμμα ε, έχει, δείχνει ευαισθησία και ενδιαφέρει ιδιαίτερα για το θέμα. Τώρα, ο εξωτερικό συναγερμό, το γεγονό, δηλαδή ότι καθίσταται δημόσια η σχετική πληροφορία και όχι μόνο ε, καταγγελωμένη προς τις αρχές αλλά και στον τύπο, εμένα μου φαίνεται ότι πρέπει να είναι ε, κάτι εξαίρεση. Να καταγγελθεί δημόσια εφόσον υπάρχει κάποιο βαρύ παράπτωμα ή εάν οι διαδικασίες εσωτερικού συναγερμού εντός της επιχείρησης δηλαδή δεν έχουν αποδώσει. Εάν δηλαδή ε, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που έχουν θεσπίσει οι επιχειρήσεις, κάποιες λειτουργούν, κάποιες όλες όχι, θα πρέπει να επαγρυπνεί κανείς. Παρ' όλα αυτά εμένουμε στην αρχή σύμφωνα με την οποία εξωτερικός ε, συναγερμός θα πρέπει να είναι κάθε εξαίρεση. Δεύτερο, για να είναι προστατευμένη αυτοί που θεωρούνται καταγγέλλοντες, θα πρέπει το φυσικό οικονομικό πρόσωπο να ε, δρά με καλή πίστη και χωρίς ίδιο συμφέρον. Θα πρέπει δηλαδή να αποκλείσουμε από το πεδίο προστασίας των καταγγελόντων αυτούς που έχουν κάποιους δικούς τους λογαριασμούς να ξεκαθαρίσουν ή που θέλουν να παρενοχλήσουν ή που ε, ε, για την περίπτωση αυτή θα καταφύγουν πίσω από το καθεστώς του καταγγέλλοντος για να προκαλέσουν προβλήματα στην επιχείρηση και ενδεχομένως να ε, βλάψουν την ε, ε, νομική ασφάλεια της επιχείρησης ή εν πάση περιπτώσει που διαθέτουν κακή πίστη. Αλλά θα πρέπει να μην έχουν ίδιο συμφέρον εάν θέλουμε το καθεστώς αυτό των καταγγελόντων να είναι νόμιμο και αποδεκτό από όλους. Τρίτη αρχή, θεωρώ ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα βεβαίω υπέρ των καταγγελόντων, αλλά και των ε, προσώπων κατά το οποίο στρέφονται οι καταγγελίε διότι υπάρχει και το τεκμήριο αθότητας και δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από τι ψευδει κατηγορίε. Βεβαίω και θα πρέπει η πληροφορία, οι πληροφορίε που πρέπει να καταγγελθούν να μπορεί να γίνει η καταγγελία αυτή, αλλά θα πρέπει ποτέ να αποβεί αυτό σε βάρος του τεκμηρίου αθότητος που είναι θεμελιώδης αρχή και όλοι στις χώρες μας. Έχουμε παραδείγματα φυσικών ή και νομικών προσώπων τα οποία κατηγορήθηκαν αδίκως και θεωρώ ότι για μας θα πρέπει η αρχή αυτή να παραμείνει θεμελιώδης και ε, να ισχύει για όλες τις πολιτικές ομάδες. Εν τέλει, σε ό,τι αφορά την επαγρύπνηση, ας μην αντιστρέψουμε καταρχήν το βάρος αποδείξεως. Να εξηγήσω. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις αρχής, όπως στην περίπτωση αντιπίνων. Θεωρώ παρόλα αυτά ότι πρώτα-πρώτα ο καταγγέλων θα πρέπει να φέρει την ευθύνη να αποδείξει το αληθές των ισχυρισμών του και όχι τόσο η επιχείρηση ή το πρόσωπο καθού στρέφεται κατηγορία να αποδείξει δηλαδή αρνητικά ότι δεν έχει πράξει αυτό για το οποίο κατηγορείται θα πρέπει να παραμείνουμε στα πλαίσια μιας υγιούς αρχής, ότι δηλαδή αυτός που ζητεί κάτι οφείλει και να αποδείξει. Είναι βασικές αρχές αυτές, είναι και θέματα συζητήσεως. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε και να συμβαστούμε από αυτόν, εν πάση περιπτώσει, και ζήτημα επί των οποίων χρειάζεται, ζητήματα μάλλον επί των οποίων χρειάζεται επαγρύπνηση. Όπως και οι άλλοι σκιώδεις θα αναζητήσω κι εγώ την αναγκαία ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη καταγγελίας παρανομιών και βεβαίως από την άλλη μεριά την ε, προστασία των προσώπων και του επιχειρηματικού απορρίτου και των επιχειρήσεων γενικότερα. Κύριε Le Και εγώ με τη σειρά μου να πω ότι χαίρομαι πολύ με το κείμενο αυτό. Ε, γιατί σημαίνει ότι η Κομισιόν εισάκουσε το Κοινοβούλιο. Ε, υπενθυμίζω ότι πρόκειται για απέτηση η οποία προέκυψε από τις συζητήσεις μας για το, το απόρριτο των ε, των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ε, έπρεπε να προσπαθήσουμε να απαλύνουμε αυτές τις, τους προβληματισμούς ε, μέσα από το κείμενο για τους καταγγέλλοντες. Χαίρομαι ε, γιατί ο νόμος, ε, ο γαλλικός νόμος της 9 η 12ου 2016 εν μέρη έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης για το κείμενο αυτό. Ε, να πούμε ότι θα είναι μάλλον από ό,τι φαίνεται αποτελεσματική η προστασία των καταγγελόντων. Προβλέπεται και προστασία για δικαιολόγητες διώξεις και βεβαίως η διαδικασία καταγγελίας ε, συμμορφούνται με αυτό που εγώ ήλπιζα, δηλαδή βασίζεται στην αρχή ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από εσωτερική διαδικασία πρώτα, πριν περάσουμε στην εξωτερική διαδικασία και που βεβαίως ε, σε περιπτώσεις ε, έκτακτης ανάγκης μπορεί κανείς να προσφύγει στην εξωτερική, επομένως την γνωστοποίηση της καταγγελίας. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όμως για κάποια σημεία. Το πρώτο είναι η αντιστροφή του βάρους της απόδειξη. Εγώ πάντα έλεγα ε, ότι δεν είμαι καθόλου υπέρ αυτής ε, της ιδέας. Είναι πολύ κακή ιδέα. Ε, θέλουμε οπωσδήποτε να προστατέψουμε τον καταγγέλλοντα και πάμε πολύ μακριά. όταν απειλείται με αντίπεινα θα πρέπει εκείνος να αποδείξει το εύρος των αντιπίνων. Επίσης δεν βλέπω πολύ θετικά το θέμα της ανωνυμίας. Ο κύριος Ντυρόν από ό,τι φαίνεται είναι αναφανδόν υπέρ. Πιστεύω ότι θα πρέπει, ε, ναι υπάρχουν περιπτώσεις ε, που πρέπει να υπάρξει ανωνυμία αλλά πιστεύω ότι είναι επικίνδυνο να ορίσουμε την ανωνυμία ως γενική αρχή. Επίσης και κάτι το οποίο εξ αρχής στη διάρκεια της συζήτησης ε, είχα αναφέρει, ε, βλέπω ε, με ιδιαίτερα θετικό μάτι την, το ιατρικό απόρριτο, προστασία ιατρικού απορρίτου, εθνικών στοιχείων απορρίτου άμυνας κτλ. Δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν να επιτρέψουμε να αποκαλύπτονται τέτοιου είδους μυστικά και απόρριτες πληροφορίες προς χάρη της καταγγελίας σε Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Να υπενθυμίσω ότι έχει σταλεί σε 13 επιτροπές ο φάκελος αυτός ε, για γνώμο δότηση, κόντε, κονέμπλε, λίμπε, αλλά Βλέπω μόνο τον κύριο Λούντβικσον που μπορεί να είναι σχετικός ε, με αυτού του είδους τις γνωμοδοτήσεις. Ε, θέλετε να πάρετε το λόγο, μα και βέβαια θέλω. Εγώ αντικαθιστώ την Γκίτελαντ. Η ομάδα μου και εγώ περιμέναμε την πρόταση αυτή εδώ και, ε, εδώ και χρόνια. Επομένως είναι πάρα πολύ καλό που επιτέλους έχουμε την πρόταση αυτή στα χέρια μας. Ωστόσο, πιστεύω ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Η πρόθεση της οδηγίας είναι η προστασία των ε, καταγγελόντων. Είναι σημαντικό ε, για τους μεμονωμένους καταγγέλλοντες να κατανοούν ε, με ευκολία πότε είναι προστατευμένοι και πότε όχι υπάρχουν ακόμα κάποιες ε, ασάφειες ε, και αβεβαιότητες. Ας πούμε, είναι λυπηρό που το άρθρο 153 δεν προτείνεται ε, ως μία από τις πολλές δομικές βάσεις που έχουν προταθεί. Και επίσης, επομένως, έτσι δεν λαμβάνονται υπόψη τα εργασιακά δικαιώματα. Επίσης, η καταγγέλλοντες ε, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί πότε ε, προχωρούν και πώς ορίζεται η εσωτερική και η εξωτερική καταγγελία. Επίσης θα πρέπει να γίνει πιο σαφής ε, ο ρόλος των συνδικάτων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 καθορίζεται ο ρόλος αυτός, αλλά πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει επιπλέον αποσαφήνιση και διευκρίνηση όσον αφορά τους διάβλους ε, των ε, συνδικαλιστικών οργανώσεων. Ε, και αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θέλει η Κομισιόν να πάρει το λόγο. Όχι, από ό,τι φαίνεται. Κυρία Ροζιέρ, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Κυρία Ροζιέρ, απλώς ε, να πούμε ότι έχουμε αρκετά φιλόδοξο χρονικό ορίζοντα ε, και θα πρέπει όλοι να κινητοποιήσουμε τις δυνάμεις μας έτσι ώστε να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε την εργασία ε, μέσα στα χρονικά πλαίσια. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν με το σημείο 20 της ημερησίας διατάξεως, ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά ε, αντιπροσωπητικές δράσεις για την προστασία συλλογικών δικαιωμάτων ε, καταναλωτών. Η συγητής είναι ο κύριος Διδιέ, Ζωφρουά Διδιέ, στον οποίο και δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρχάς για την συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η οποία έχει σαν στόχο την καλύτερη προστασία των καταναλωτών. Το σχέδιο αυτό οδηγίας έχει σαν βασικό στόχο τον εξυγχρονισμό την οδηγία επιβολής του 2009, εγγράφεται στα πλαίσια του σχεδίου πρωτοβουλίας του ε, ΛΕΝΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 12 και ανταποκρίνεται σε μια πραγματική ανάγκη γιατί εννέα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν πάντα εισάγει μηχανισμούς συλλογικής αποζημίωσης. Υπάρχει λοιπόν μια πολυδιάσπαση των εθνικών νομοθεσιών εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εις βάρος συνεπώς των καταναλωτών. Ποιος είναι ο στόχος μας. Θέλουμε να προσπαθήσουμε από κοινού μαζί με τους σκιώδεις εισηγητές, μαζί και με την Επιτροπή ΙΝΚΟ, να βρούμε μία απαραίτητη ισορροπία ανάμεσα στην αυξημένη προστασία των καταναλωτών και στην νομική ασφάλεια των επιχειρήσεων. Δηλαδή ανάμεσα στη μία στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη, έτσι ώστε να αποζημιούνται η βλάβη, και κυρίως για να αποφύγουμε νέες παραβιάσεις του ευρωπαϊκού δικαίου, θα πρέπει να έχουμε και στόχους αποτροπής και όχι μόνο διορθωτικούς θεραπευτικούς. Να δίνουμε λοιπόν εγγυήσει ε, και για τις ε, καταχρηστικές προσφυγές. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν τις επόμενες εβδομάδες να εργαστούμε πάνω σε πολλά θέματα μαζί και θα ήθελα να ξεκινήσω με κάποια πρόταση μιας σκέψης. Το πρώτο είναι το πεδίο εφαρμογής. Εδώ το σχέδιο οδηγίας καλύπτει πολλαπλούς τομείς που μπορεί να ε, έχουν, να χαρακτηρίζονται από το από τη συλλογική προσφυγή, τουρισμός, εστίαση και θα πρέπει εδώ να προσπαθήσουμε να δούμε αν θα πρέπει να διευρύνουμε το πεδίο αυτό εφαρμογής. Δεύτερον, ένα άλλο σημείο συζήτησης. Ποιοι έχουν δικαίωμα να ασκήσουν τέτοιου προσφυγές. Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια σήμερα τα οποία λαμβάνονται υπόψη στην πρόταση οδηγίας. Ε, Καλής φήμης καταρχάς. Θα πρέπει ε, να μην έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, η χρηματοδότηση να είναι διαφανής, ε, το συμφέρον της αποδείξιμο. και μόνο οι ανεξάρτητοι οργανισμοί εκπροσώπησης των καταναλωτών να έχουν αυτή την δυνατότητα. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε πλήρως τα κριτήρια αυτά για να μπορέσουμε να εναρμονίσουμε την νομοθεσία. Αυτός είναι ο βασικός στόχος. Και θα πρέπει επίσης ε, να θέσουμε και το εξής ερώτημα της, ε, του θεμητού ή μη, αν θέλετε, της νομιμοποίησης ή μη αυτών των οντοτήτων. Ένα τρίτο θέμα αφορά στην ενημέρωση και στο εύρος της ενημέρωσης των καταναλωτών. Το σχέδιο οδηγίας θα πρέπει να καθορίσει καλύτερα, σαν παράδειγμα, αν όλοι οι α, καταναλωτές εμπλέκονται στην δικαστική διαδικασία ή αν θεωρούμε ότι τα φυσικά οι νομικά πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν δεν μπορούν να το κάνουν παρά μόνο εθελοντικά. Και τέλος ένα τελευταίο σημείο συζήτησης, σημαντικό σημείο συζήτησης, αν και ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός, αφορά τους κινδύνους παραβιάσεων, παραβάσεων διασυνοριακών σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι κάνουμε εδώ, κάνουμε μία δίκη αναχώρα ή μία δίκη ενιαία για το σύνολο της Ένωσης. Και αν θεωρήσουμε ότι θα πρέπει να γίνεται σε κλίμακα ευρωπαϊκή, με ποιο κριτήριο θα επιλέγουμε την δικαιοδοσία. Θέλουμε να εναρμονίσουμε ή να αφήσουμε κάθε χώρα να διευκρινίσει η να αφησουμε καθε χωρα να διευκρινισει ιδια το πεδίο εφαρμογής της. Και εδώ τίθεται το θέμα του ανταγωνισμού των δικαιοδησιών, ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής, ανάλογα με το βάρος της ποινή, ανάλογα με την ύπαρξη ή μη μίας Οντότητα που να έχει το δικαίωμα να κάνει την προσφυγή. Συνεπώς λοιπόν βλέπουμε ποια είναι τα σημεία συζήτησης, ε, τα καταγράφουμε, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε με τις πολιτικές ομάδες. Η δική μου φιλοσοφία δράσης είναι απλή, να προσπαθήσουμε να βρούμε, αν θέλετε, μια σωστή ισορροπία, έτσι ώστε να προστατεύσουμε τους καταναλωτές καλύτερα. Αυτό είναι αναμενόμενο, είτε είναι πελάτες, αγοραστές, ταξιδιώτες, επενδυτές. Και από την άλλη θα πρέπει, και αυτός είναι ρόλος μας, να μπορέσουμε να προσφέρουμε εγγυήσεις επαρκής για τις επιχειρήσεις οι οποίες ανησυχούν για το επίπεδο νομικής ασφάλειας και για τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους. Αν μπορέσουμε να βρούμε αυτήν την ισορροπία, η οποία θα απαιτήσει πολλά από μας και αυτό είναι και το πνεύμα του Κοινοβουλίου, ε, μια προσπάθεια ε, δημιουργίας συνένεσης, συμβιβασμών, θα καταλήξουμε νομίζω σε ένα πλήρες ε, κείμενο, μια πρόταση αρκετά πλήρη, έτσι ώστε και στα πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας να δείξουμε ότι η Ευρώπη χρησιμεύει, εν να προστατεύει τους καταναλωτές και να βοηθά την αποζημίωσή τους. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε αξιόπιστοι θα πρέπει να παράσχουμε την κατάλληλη νομική προστασία και ασφάλεια ε, για τους καταναλωτές που δεν θα πρέπει να πέφτουν θύματα σε κοινοτικό επίπεδο. Τώρα, ε, τις επόμενες μέρες ε, θα καθορίσω τον χρονισμό της διαδικασίας, του Ίτερ που ακολουθούμε. Δύο είναι οι στόχοι. Ο πρώτος είναι να προχωρήσουμε με ταχύτητα και ο δεύτερος, όπως και να έχουν τα πράγματα, η οδηγία αυτή θα πρέπει να γίνει δεκτή στην Ολομέλεια πριν το τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου. γιατί οι καταναλωτές έχουν ανάγκη από περισσότερη προστασία και εμείς οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να δείξουμε, έχουμε ανάγκη να δείξουμε τους επόμενους μήνες σε ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι πράγματι ασπίδα προστασίας. Εσείς κύριε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ λοιπόν να χαιρετήσω την πρόταση την οποία μας υποβάλλει επιτέλους θα έλεγα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί η έκθεση πρωτοβουλίας είναι του 2012 είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη πρόταση και απαραίτητη πρόταση. Δεν θα επαναλάβω όλα τα επιχειρήματα τα οποία ήδη παρουσίασε ο εισηγητής. Πάντως σημειώνω εδώ την εξαιρετική επιφυλακτικότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι στα κράτη-μέλη. Φροντίζει έτσι ώστε να μην παρεμβαίνει στις αρμοδιότητες και το, ουσιώδε το ουσιώδες δίκαιο δεν φύγεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οι διαδικασίες και οι νομικές εθνικές ρυθμίσεις γίνονται πάντα σεβαστές και αν κατάλαβα καλά ε, υπάρχουν κάποια περιθώρια πλέον. Τα κρατη είναι αυτά τα οποία ορίζουν τις οντότητες που έχουν την δυνατότητα να προχωρήσουν σε προσφυγές συλλογικού τύπου. η αλλαγή στους καταλόγους ανήκει στα κρατημέλη, ο έλεγχος των χρηματοδοτήσεων παραμένει πάντα στις αρμοδιότητες των κρατών μελών και νομίζω ότι έχουμε εδώ με, ε, εξ αυτού πολλές πιθανότητες επιτυχίας. Κάποια σημεία όμως μπορεί να τύχουν βελτίωσης. Βασικός στόχος είναι ένα κράτος μέλος ας πούμε, το οποίο έχει ρυθμίσεις εθνικές πιο προστατευτικές από αυτές που κάνουμε εμείς, οι ρυθμίσεις αυτές οι εθνικές να μην αμφισβητούνται να μην αμφισβητηθούν. Πρόκειται δηλαδή για μια κατελάχιστον μορφή εναρμονισμού. Σε σχέση τώρα με το πεδίο εφαρμογής, το άρθρο 2 δηλαδή, παραπέμπει σε ένα παράρτημα το οποίο θα μπορούσαμε να επιμικίνουμε. Έχω όμως ένα ερώτημα παρατηρώ το θέμα της προστασίας των δεδομένων στο παράρτημα αυτό. Αυτό σημαίνει ότι η ηθική βλάβη θα καλυφθεί και αυτή ή μήπω θα περιοριστούμε ε, στην ηλική και μόνο βλάβη. Είναι ένα θέμα το οποίο τίθεται και χρήζει απάντηση. Σχετικά τώρα με το πεδίο εφαρμογή να πω ότι εξεπλάγει ελαφρώ γιατί βλέπω στη ρήτρα αναθεώρηση αυτό 18 παράγραφος 2 ότι το δικαίωμα των επιβατών περιλαμβάνεται στη ρήτρα αναθεώρησης. Ε, διαρωτώ με εδώ, γιατί θέλουμε να θέσουμε σε αμφισβήτηση τα δικαιώματα των, των επιβατών. Είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν με ανησυχεί, αλλά σίγουρα μου προκαλεί περιέργεια. Σχετικά τώρα με το άρθρο 6 παράγραφος 2, η απόκληση για τις λεγόμενες περίπλοκες υποθέσεις. Και εδώ θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει ορισμένες διευθυνήσεις. Αν αφήσουμε πάρα πολλά κοινά, πάρα πολλά κενά, συγγνώμη, παραθυράκια και ο ορισμός του περίπλοκου μιας υπόθεσης είναι δύσκολος. Αν και ε, εδώ αναφέρεστε ίσως το θέμα της ποσοτικοποίησης του ύψους της βλάβης. Το πέμπτο σημείο και εδώ θα ήθελα να υπάρξουν ορισμένες διευκρινήσεις. Πρόκειται για το άρθρο 16 σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές διασυνοριακές δράσεις. Εδώ εγώ θα μπορούσα να σκεφτώ μια αντιπροσωπευτική ευρωπαϊκού τύπου δράση, αλλά αυτό είναι ένα όνειρο απατηλό. Ας είμαστε λοιπόν ρεαλιστές, αλλά ας διευκρινίσουμε λίγο καλύτερα το συγκεκριμένο πλαίσιο. Κλείνοντας, Άκουσα πολλούς φόβους, επιφυλάξεις ε, για την καταχρηστική ε, προσφυγή. Νομίζω ότι υπάρχουν ρήτρες προστασίας έτσι ώστε ο φόβος αυτός να μην είναι τεκμηριωμένος. Να αναφερθώ σε κάποιες τέτοιες ρήτρες προστασίας. Σαν παράδειγμα, η ποιοτική αξιολόγηση των οντοτήτων που έχουν την δυνατότητα. Η εκκίνηση της διαδικασίας μετά από δικαστική απόφαση που διαπιστώνει την παραβίαση του δικαίου. Επίσης, ε, η διαφάνεια της χρηματοδότησης ε, της συγκεκριμένης οργάνωσης, όπως επίσης ε, και έλεγχος των συμφερόντων τρίτων. Νομίζω ότι με όλες αυτές τις απαντήσεις που δίδονται στις επιφυλάξεις και στους φόβους αυτούς, ελπίζω να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με ταχύτητα και να προσφέρουμε στον Ευρωπαίο καταναλωτή απλοποιημένες διαδικασίες, ιδιαίτερα στις εννέα χώρες, χώρες οι οποίες δεν έχουν νομοθετικές ρυθμίσεις ε, για την προστασία των των... του δικαιώματος των καταναλωτών σε συλλογική προσφυγή. Ευχαριστώ τους εισηγητές, ευχαριστώ τον εισηγητή μάλλον και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εξηγήσεις. Ja, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για τις σαφέστατες κατευθύνσεις που δώσατε. Όπως η κυρία Ντελβό και εγώ χαίρομαι πολύ, διότι έτοιμα που προβάλλουμε από πολλά χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταλήγει επιτέλους να περιληφθεί σε νομοθετική πρόταση η οποία νομοθετική πρόταση θα επιτρέψει πρόοδο διότι σιγά σιγά είναι αναγκαίο σε μια Ευρώπη που ολοκληρώνεται όλο και περισσότερο, ενοποιείται όλο και περισσότερο, δημιουργείται ενιαία αγορά και είναι σωστό να υπάρξει προστασία των καταναλωτών στην ενιαία αγορά. Διότι έχουμε αυτές τις περιπτώσεις Dieselgate, και άλλες σχετικές υποθέσεις που δείχνουν ότι είναι αναγκαίο να δώσουμε κάποια εργαλεία, κάποια όπλα στις καταναλώτριες και στους καταναλωτές που να τους βοηθούν να λύσουν προβλήματα και να μην είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Ορισμένα από αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κρίνω πολύ θετικά. Αφενός τα συστήματα που έχει προβλέψει για να αποτρέψει να δημιουργηθεί ένα νέο business model αγωγών με την έννοια ότι μη κυβερνητικέ οργανώσεις οι οποίες δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα αυτές λαμβάνουν το δικαίωμα αυτό και όχι άλλες, κάποιες άλλες. Αυτό βρίσκω σωστό και είναι σωστό να επιμείνουμε σε αυτό έστω και αν έχω δεχτεί διαβήματα από διαφόρους ε, δικηγόρους για να ρωτήσουν και γιατί όχι εμείς χρειάζεται προσοχή και νομίζω ότι ειδικά αυτό που προτείνει εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι καλό, είναι θετικό. Όπως άλλωστε και η κυρία Ντελβό, θεωρώ και εγώ ότι είναι ισορροπημένη η πρόταση και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε και μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να δώσουμε αυτονομία και να αφήσουμε μάλλον αυτονομία και κυριαρχία στις χώρες μέλη, ώστε να έχουμε και τη δυνατότητα πραγματικά να περάσει τελικά η νομοθεσία, διότι γνωρίζουμε ότι ο πολιτισμός, η κουλτούρα ας πούμε, της νομολογίας διάφορες χώρες μέλη είναι διαφορετική. Και βεβαίω οι παραδόσει είναι διαφορετικέ και οφείλουν να τηρηθούν. Και είναι σωστό επίση που το πεδίο εφαρμογή περιλαμβάνει 59 οδηγίε και κανονισμού επαρκή αριθμό. Θα κάνω κάποιε προτάσεις, κάποιε τροπολογίε για να διευρύνω έτσι περαιτέρω το πεδίο αυτό διότι θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη να ρυθμιστούν πράγματα νομοθετικά, όπως η προσφορά ψηφιακών περιεχομένων ή δικτυακών περιεχομένων και ούτω καθεξής που ακόμα βρίσκονται στην νομοθεσία, αλλά θα πρέπει προληπτικά να τα περιλάβουμε στο πεδίο εφαρμογής, ώστε να μπορέσουν και αυτά να αντιμετωπιστούν. Έχουμε κάποιες δυνατότητες εκεί να το διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής. Πρόσεξα και εγώ το άρθρο 8 με την εξαίρεση για δικαιώματα των επιβατών. Και εγώ εξεπλάγει, όπως η κυρία Ντελβό. Χρειάζεται λοιπόν να εξετάσει κανείς εδώ ε, τι κρύβεται από πίσω και να αποφευθεί το ενδεχόμενο να παρισφρήσει κάποια ανασφάλεια δικαίου λόγω των περίπλοκων ρυθμίσεων. Ίσως εκεί μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί με την διάταξη αυτή. Εγώ πάντως δεν κατάλαβα για ποιο λόγο κάνει τη σχετική πρόταση. Εν τέλει πάντως θέλω να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα για την πρόταση που έχουμε λάβει και όπως ο κύριος Ντιντιέ και η κυρία Ντελβό θεωρώ ότι η πρόταση μπορεί με να βελτιωθεί, στο σύνολό της όμως είναι καταρχήν θετική και ε, θα πρέπει όντως να την επεξεργαστούμε περαιτέρω. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Έχω και εγώ ένα σχόλιο. Στην εκλογική μου περιφέρεια, η πρόταση της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηλαδή, έχει γύρει ενδιαφέρον και θα έλεγα και συγκρατημένη αισιοδοξία. Και το βασικό ερώτημα που άκουσα και ακούω είναι η βασική ανησυχία να διασφαλίσουμε ότι το σύστημα δεν θα μπορεί να γίνει αντικείμενο κατάχρησης όπως γίνονται οι συλλογικές αγωγές αποζημίωσης στις ΗΠΑ. Το ερώτημα αυτό πιστεύω θα ακούγεται διαρκώς σε όλη τη διάρκεια δηλαδή της νομοθετικής διαδικασίας. Επιθυμεί τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει το λόγο. Ορίστε κυρία μου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές, εισηγητής, συνεισηγητές και εσάς κύριε Πρόεδρε για την υποδοχή που επιφυλάξατε στην ε, πρόταση. Ευχαριστώ και για την εισαγωγή, πλήρη εισαγωγή που κάνατε και δείχνει πραγματικά σε βάθος κατανόηση της προτάσεώς μας που εν πάση περιπτώσει είναι αρκετά περίπλοκη και τα λόγια σας είναι πολύ ενθαρρυντικά για μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχω κάποια πληροφοριακά στοιχεία που μπορώ να προσθέσω σε σχέση με κάποια τμήματα της οδηγίας που συζητήθηκαν μέχρι τώρα από τον εισηγητή και τις συνεισηγητρίες σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή. Ορθώς κατανοήσατε ότι εμείς προβλέπουμε να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογή της τρέχουσας οδηγίας για να περιλάβουμε παραβιάσεις του δικαίου προστασίας καταναλωτών για να περιλάβουμε και κάποιους μηχανισμούς του κοινοτικού δικαίου σε πλήρωνες τομείς όπως μεταφορές, περιβάλλον, ενέργεια, υγεία που περιέχουν όμως και διατάξεις για τις σχέσεις μεταξύ εμπόρων και καταναλωτών και τα σχετικά δικαιώματα εκαθέρωθεν. Και συζητούμε επίση το ενδεχόμενο να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή και ο λόγος για τον οποίο, για να καθαρό ο λόγο για τον οποίο επιλέχθηκαν αυτά τα εργαλεία. Ειδικότερα τώρα για τα δικαιώματα των επιβατών εναρίων μεταφορών και σιδηροδρομικών μεταφορών. Γνωρίζετε ότι συζητείται πρόταση και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο για τα δικαιώματα των επιβατών σε αυτούς τους τομείς μεταφορών. Στη δική μας πρόταση περιέχονται στοιχεία για να δοθεί η δυνατότητα στους καταναλωτές να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και ατομικά για αποζημιώσεις όταν έχει σημειωθεί παραβίαση. Και η επιθυμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν να δούμε πώς θα προχωρήσουν οι προτάσεις αυτές και η πρόταση αυτή και όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισής της να δοθεί στους καταναλωτές επαρκής, επαρκής προστασία στο διμερές επίπεδο, ατομικά δηλαδή και όχι σε αυτά τα πλαίσια της συλλογικής αποζημίωσης, collective redress. Αυτός είναι ο στόχος της ε, αναθεώρησης που προτείνουμε στο άρθρο 18 της, ε, του σχεδίου οδηγίας μας. Βεβαίως, να συζητήσουμε μαζί σας και να σας δώσουμε και άλλα συμπληρωματικά στοιχεία. Σε ό,τι αφορά τις ε, οντότητες που έχουν το δικαίωμα που απορρέει από την οδηγία, έχουμε περιλάβει κάποια κριτήρια. Ρωτάτε γιατί τα κριτήρια αυτά. Σε ό,τι αφορά τους τύπους αυτού οντοτήτων. Ο στόχος μας δεν είναι να προσφέρουμε μονοπόλιο σε οργανώσεις καταναλωτών και στις αρχές προστασίας καταναλωτών. Ο στόχος μας είναι περισσότερο να δείξουμε ότι οι χώρες μέλη οφείλουν εν πάση περιπτώσει εφόσον οι σχετικές οργανώσεις πληρούν τα κριτήρια να είναι οι ειδικέ αυτές ε, οργανώσει οι οποίες θα έχουν, οι οντότητες δηλαδή, οι οποίες θα έχουν, οι φορείς αν θέλετε, που θα έχουν αυτά τα δικαιώματα. Τι γίνεται τώρα, μάλλον η κυρία Ντελβό αναφέρθηκε στο άρθρο 1 παράγραφος 2. Τι γίνεται εάν οι χώρες μέλη έχουν τέτοια συστήματα τα οποία λειτουργούν καλά. Αυτό που λέει το άρθρο 1 παράγραφος 2 είναι ότι οι χώρες μπορούν να διατηρήσουν τα εναλλακτικά του συστήματα τα οποία επίσης έχουν ως στόχο την προστασία των συλλογικών δικαιωμάτων των καταναλωτών. Θα μπορούσε λοιπόν να μιλήσει κανείς για ελάχιστη εναρμόνιση. Ήδη έχουμε συζητήσει πολύ βεβαίως με το Συμβούλιο για το άρθρο αυτό από τότε που καταθέσαμε την πρόταση προχωρώντας τις εργασίες μας θα δούμε αν πρέπει να διευκρινιστεί περισσότερο το περιεχόμενο του σχετικού άρθρου. Αυτό είναι ζήτημα που πρέπει να συζητηθεί. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, κύριε Συγητά και κύριε Συνεισηγήτρες, αυτά είναι κάποια πληροφοριακά, πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία. Είμαστε, είμαστε εννοείται στην διάθεσή σας για να συζητήσουμε οποιαδήποτε θέματα σας απασχολούν σχετικά με την οδηγία. Thank you very much. Mr. Uh, wanted to take... Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Βόνκεβαλτ. Ευχαριστώ. Συμπληρωματική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εγώ εκφράζω τη χαρά μου για την πρόταση. Και θεωρώ ότι και οι safeguards, τα εχέγγυα που έχουμε περιλάβει για να μην υπάρξει κατάχρηση αυτού του δικαιώματος αγωγής, στη συλλογική αγωγή θα πρέπει να επεκταθεί αυτή και σε παροχές. Εφόσον υπάρξει αγωγή σχετική με παροχές από οργάνωση καταναλωτών, αυτό για μένα είναι κάπως ε, δύσκολο, κάπως περίπλοκο. Εάν τώρα ζητήσει μια παροχή, μια οργάνωση καταναλωτών, για παράδειγμα καταβολή μιας αποζημιώσεως, ποια θα είναι τότε συγκεκριμένη παροχή θα γίνει προς την οργάνωση καταναλωτών θα δοθεί σε κάποιον ο οποίος έχει καταχωριστεί σε ένα μητρό αλλά δεν είναι ενάγων ε, ίσως δεν έχω αρκετή φαντασία για να ε, αντιληφθώ όλο το νόημα και μου χρειάζεται ίσως κάποια διευκρίνηση. Η Κομισιόν θέλει να απαντήσει μήπως. ίσως ε, να δώσω κάποια στοιχεία απάντησης. Δεν προτείνουμε ε, να ρυθμίσουμε τον ε, βασικό νόμο, τον ουσιαστικό νόμο. Η απάντησή μου ε, η απάντησή μου λοιπόν είναι θα εξαρτηθεί από ε, ποια, ε, από ποιο τομέα ας πούμε, στο ποιο τομέα υπάρχει παραβίαση, αλλά εντάξει μπορώ κάποια στιγμή να σας δώσω περαιτέρω πληροφορίες. Δεν ξέρω αν η εισηγήτρια θέλει, ο εισηγητής θέλει να κάνει κάποια σχόλια, όχι. Να συνεχίσουμε λοιπόν με το σημείο 21, ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά ε, την ε, γρήγορη επίλυση ε, και εμπορικών διαφωνιών και το λόγο έχει ο Ταντέος Ζουιφκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εδώ θα έχουμε μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό, γιατί σήμερα ξεκινούμε την εργασία μας ε, για αυτή την πρόταση ε, πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου για ε, επιταχυμένες διαδικασίες επίλυσης εμπορικών διαφωνιών. Ο στόχος είναι να βρούμε κάποια νέα στοιχεία για τη διευκόλυνση τη ενιαίας αγοράς. Αυτό, ένα τέτοιο εργαλείο λοιπόν είναι απαραίτητο και νομίζω ότι πρέπει να είναι σαφής η απάντηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουμε στην διάθεσή μας και λαμβάνοντας υπόψη και τις εκτιμήσεις ε, της Παγκόσμιας Τράπεζας, η λύση των διασυνοριακών ε, εμπορικών ε, διαφορών ε, είναι διαδικασία μακρά και σε ορισμένες χώρες μπορεί να κρατήσει μέχρι και πέντε χρόνια τα μέρη τα οποία εμπλέκονται σε αυτήν την ε, διαφορά, σε αυτή την διαμάχη ε, μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολύ περίπλοκα εργασία, ε, εργαλεία συγγνώμη, και πολύ συχνά γίνεται αναφορά και σε άλλο δίκαιο κτλ. Δεν υπάρχει λοιπόν Μπορεί να υπάρξει δηλαδή νομική ασφάλεια και επομένως καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα τα οποία μπορούν να προκύψουν μπορεί να είναι πολύ σημαντικά ε, και σε ορισμένες περιπτώσεις ε, μπορεί να σημαίνουν ε, ότι θα σταματήσουν ας πούμε οι χρηματοδοτήσεις και ε, ενδεχομένως ε, η περιού ο λόγος χρηματοδοτήσεις μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικές για την λειτουργία και την επιβίωση της ε, επιχείρησης. Στη διάρκεια της αναθεώρησης του κανονισμού Βρυξέλλες 1 καταφέραμε να απλουστεύσουμε και να βελτιώσουμε σημαντικά τα θέματα τα οποία σχετίζονται με την ε, νομολογία όσον αφορά τις ε, αποφάσεις ε, αστικές και εμπορικές. και γενικώ οι αποφάσεις που έχουμε πάρει, καθώς επίσης και τα σχετικά νομοθετικά κείμενα, είχαν καλή ε, είχαν ε, καλή ε, επίπτωση. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα άλλο θέμα. Αναφέρομαι στις ελάσσονος σημασίας διαφορές και την επίλυσή τους. Ας πούμε προσφυγές καταναλωτών ή ε, οι προσφυγές οι οποίες αφορούν ποσά χαμηλότερα από τις 5.000 ευρώ. Και αυτό είναι ένα θετικό βήμα το οποίο θετικώς δέχτηκαν και οι πολίτες της Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, όσον αφορά λοιπόν ε, και απέναντι σε αυτά τα συγκεκριμένα θέματα, πιστεύω ότι μπορούμε να στραφούμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να παρουσιάσουμε νομοθετική, νομοθετικό ε, κείμενο για, τις, ε, ε, για την επίλυση διασυνοριακών διαφορών, κυρίως όσον αφορά τις σχέσεις B2B, business to business δηλαδή. Ε, υπάρχει και μία διαδικασία που μπορούμε να την ονομάσουμε αστική ευρωπαϊκή επιταχυμένη διαδικασία ε, θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να επιταχυνθούν αυτές ε, οι διαδικασίες οι οποίες όπως είπα και προηγουμένως μπορεί να διαρκέσουν πάρα πολλά χρόνια. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι θα πρέπει να είμαστε σε θέση να μειώσουμε τις διαδικασίες αυτές σε μια χρονική περίοδο έξι μηνών και πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό θα βελτιώσουμε πάρα πολύ τις διαδικασίες. Αλλά βεβαίως ε, αυτό αφορά ε, και θέματα όπως είναι η ασφάλεια δικαίου όπως είναι η δυνατότητα να συνεχίσουν τις εργασίες τους οι επιχειρήσεις, μείωση του κόστους κλπ. Επίσης, έχουμε τον κανονισμό ε, Ρώμα 1 ε, όσον αφορά τις συμβατικές υποχρεώσεις. Αλλά πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επιλογής του κατάλληλου ε, της κατάλληλης νομικής ε, βάσης και όσον αφορά τον εφαρμοσματικό νόμο αυτός δεν σχετίζεται απαραίτητα με την έδρα της επιχείρησης ή δεν συνδέεται άμεσα και αποκλειστικά με ένα συγκεκριμένο με μια συγκεκριμένη σύμβαση. Αυτή η επιταχυμένη διαδικασία ε, με κανένα τρόπο δεν θα ε, μπορούσε να αποτελέσει πρόσκομα στις διαδικασίες που προβλέπονται ε, στο Ρώμη 1. Πρόκειται για ένα συμπληρωματικό εργαλείο που διασυνδέει την επιλογή του εφαρμοστέου κειμένου και την ε, ε, έδρα της εταιρείας ή ε, την χώρα στην οποία εκτελείται το συμβόλαιο. Σύμφωνα, σύντομα θα βγει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ε, συνεργασίες μεταξύ των διαφόρων ε, επιχειρήσεων ε, και μάλιστα σε διασυνοριακό επίπεδο είναι όλο και πιο έντονες και επομένως είναι καλό να έχουμε ένα εργαλείο καινούριο, είναι σκόπιμο και δόκιμο να έχουμε ένα καινούριο εργαλείο που θα διευκολύνει τις ε, ε, σχέσεις. Ε, αυτή είναι η πρώτη φορά που συζητούμε το θέμα. Καλό θα ήταν να ακούσω κάποιες απόψεις, να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων έτσι ώστε να δούμε ακριβώς με ποιο τρόπο μπορούμε να συμβάλλουμε στη συζήτηση αυτή κατά την έννοια αυτή βεβαίως πολύ σημαντική και σίγουρα θα συμβάλλει και η αυριανή ακρόαση Δεν νομίζω ότι έχω τίποτα άλλο να σας πω. Ζητώ από τους συναδέλφους ε, να ε, παρουσιάσουν την άποψή τους έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ντελβό. Ευχαριστώ. Και έπρεπε να φύγει εκτάκτος στην Ιταλία. Θα διαβάσω το σύντομο μήνυμά του. Θέλω να ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω κάποια σύντομα προκαταρτικά σχόλια, μιας και η συζήτηση μόλις έχει ξεκινήσει και το των εργασιών. Αυτό το οποίο όμως μπορώ να πω είναι να υπογραμμίσω κάτι το οποίο προφανώς άπτεται τίκο. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι για τις μη νομοθετικές πρωτοβουλίες, τις οποίες γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, υπάρχει θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι για τις μη νομοθετικές πρωτοβουλίες, τις οποίες γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, υπάρχει της δικαιοσύνης. Συνεπώς λοιπόν έχουμε έναν τομέα εδώ όπου κάτι μένει να γίνει και θα παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλη ενδιαφέρον την πρόοδο της ε, συγκεκριμένης έκθεσης. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν βλέπω κάποιο άλλο σχόλιο. Ο εισηγητής έχει εκ νέου το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους για τα αρχικά σας συντροπολογιών, 69 στο σύνολό τους. για ε, τις διεκδικήσεις των τρίτων μερών. Θέλω να ευχαριστήσω τους... Ε, We don't always solve them in the same way. Ε, there are three Υπάρχουν λοιπόν τρία σημεία τα οποία θέλω να θέσω. Το ένα ε, σχετικά με τον κανονισμό Ρώμη 1. Δεύτερον, χρονοδιάγραμμα για τον καθορισμό της νόμιμης κατοικίας το θέμα τίθεται σε πολλές τροπολογίες, όπως την 24. Στην έκθεσή μου εγώ προσπάθησα να βρω κάποιες λύσεις, εξαιρώντας κάποιους τομείς από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, στα πλαίσια του άρθρου 14 παράγραφου θέση, ότι ε, μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στην περίπτωση συμβατικού τύπου ε, και όχι μη συμβατικού ε, τύπου διεκδικήσεων. Συνεπώς, δεύτερον, ο χρόνος... Ε, the point I wanted to make is that ε, this... της συνήθους κατοικίας του, των εμπλεκομένων. Αυτό τίθεται σε περιπτώσεις όπου ένας οικονομικός οργανισμός και ε, τρίτον σε θέματα προστασίας των καταναλωτών. Εδώ ζητάμε για μια ενισχυμένη προστασία καταναλωτή στην πρόταση. Προσπάθησα να αντιμετωπίσω το θέμα αυτό και στη δική μου έκθεση στην τροπολογία 14. Τροπολογία τίθεται σαν θέμα. Appropriate Λοιπόν, αυτά είναι κάποια παραδείγματα τα οποία σας έδωσα τώρα σημείων στα οποία νομίζω ότι έχουμε μια κοινότητα ανησυχιών. κυρία Ντελβό έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω καταρχάς να σας ευχαριστήσω ως εισηγητή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βοήθεια και την εξηγήσει σε ένα θέμα ιδιαίτερος τεχνικό. Ε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Στόχος του κειμένου είναι ξεκάθαρος. Θέλουμε μεγαλύτερη νομική ασφάλεια. Και δεν βλέπω εδώ την ανάγκη να υπάρξει μία εξαίρεση για τυπλοποιήσεις. Δεν ξέρω ε, αν θα πρέπει πράγματι να υπάρξει μια ξεχωριστή μεταχείριση των μεγάλων πιστοτικών ιδρυμάτων. Εγώ δεν έχω πάρει μια ικανοποιητική απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα. Και επίσης από κοινού με την κυρία Γκέφαρτ έχουμε προσπαθήσει, θελήσαμε να διευκρινίσουμε ότι σε περιπτώσεις όπου εμπλέκονται οι καταναλωτές, οι περιπτώσεις αυτές θα καλύπτονται έτσι και αλλιώς από το δίκαιο της κατανάλωσης και την προστασία των καταναλωτών. Αλλά παρόλα αυτά είμαι βεβαία ότι θα μπορέσετε να μας οδηγήσετε σε μια σωστή θέση της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ η κυρία Γκέπχαρτ. Ε, να εξασφαλιστούν τα δικαιώματά τους Στι χώρε μέλη. Δεν έχουμε το ίδιο δίκαιο σε πολλά ζητήματα σε όλες τις χώρε μέλη. Θα χρειαστεί να προσέξουμε ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε, καθώς και την... τον εισηγητή. Ναι, ναι, τα σημαντικότερα σημεία για την σχέση με τη Ρωμιένα, για την Για την ε, σχέση με τη Ρώμη 1 υπάρχουν διαφορετικέ απόψει ενδεχομένω ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή τη Ρώμη 1 και το δικό εφαρμοστέο δίκαιο και για δικαιώματα in personam, προσωπικά, που μπορούν να απαιτηθούν απέναντι σε κάποιον ο οποίο δεν σέβεται τι υποχρεώσει του. Ενώ στην παρούσα πρόταση μιλούμε για δικαιώματα in rem, δηλαδή έργα όμνε που μπορεί να περιλαμβάνουν και ακόμη και τον οφειλέτη. Υποκείμενα. Ε, θα βρούμε νομίζω εν τέλει κοινό ε, έδαφος στο περιφαρμογή των δύο κανονισμών. Για... Όταν χρησιμοποιούμε την φράση material time στην πρόταση, αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί και να λάβει την πρόταση της ε, υποχρεώσεις της Ρώμης 1 και τελικώς θα αποφασίσει το, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Για να, να δίνει και ποιος θα είναι ο πραγματικός χρόνος για την σύναψη της ε, σύμβασης, κάτι που οι νομοθέτες θα συζητήσουν μεταξύ τους και εμείς θα είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσουμε. Για την προστασία του καταναλωτού, η Κομισιόν δεν τα ανταποκρινόμαστε στην επιθυμία του Κοινοβουλίου να μην θυγούν υποχρεωτικές διατάξεις για την προστασία των καταναλωτών. Συμφωνούμε απολύτως να καταστεί αυτό κάπου σαφές, ότι δηλαδή η πρόταση αυτή είναι υπό την επιφύλαξη των ε, ε, δικαιωμάτων των καταναλωτών. Έχει τεθεί και που ανέφερε η Αντελβό είναι λύση για τις ασφάλειες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια συμβαστική λύση στην πρόταση που θα μπορούσε να καλύψει ισχύ το δίκαιο του Ασάινορ στην ε, χώρα μέλος κατοικίας και να σας πω ότι 10 Ιουλίου προβλέπεται η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας. Ωραία, συνεχίζουμε. και να σας πω ότι 10 Ιουλίου προβλέπεται η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας. Ωραία, συνεχίζουμε με το σημείο 23. Θα μελετήσουμε λοιπόν την γνωμοδότευση με θέμα η πιθάσευση της παγκοσμιοποίησης ε, και τις, οι εμπορικές πτυχές της, ε, Πρόεδρε η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου πράγματι αποφάσισε ότι θέλει να ε, σκεφτεί λίγο το θέμα της παγκοσμιοποίησης, κυρίως δε τις εμπορικές πτυχές της. Ε, ε, και φυσικά δεν μπορούσε να παραμείνει σιωπηλή και η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων γιατί υπάρχει νομική πλησίαση του θέματος. Εδώ λοιπόν αναφέρω κάποιες ε, γενικές ιδέες. Πρώτη ιδέα είναι ότι η παγκοσμιοποίηση είναι μια πραγματικότητα να επαναληφθεί ε, ο σεβασμός διαφόρων αρχών, δηλαδή της εθνικής ταυτότητας και της επικουρικότητας καθώς ιδιοκτησίας ε, και είναι πολύ ευτυχή η συγκυρία που παρουσιάζω την έκθεσή μου, την γνωμοδότησή μου, συγγνώμη, με αυτήν σήμερα που μιλήσαμε για γεωγραφικών, των προστατευμένων γεωγραφικών ενδείξεων πολλές ευρωπαϊκές χώρες ε, ε, είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένες με ε, πολύ περισσότερες τέτοιες προστατευόμενες γεωγραφικές ονομασίες και ότι στις μελλοντικές αφορά επενδύσεις είναι επενδύσεις ε, συνδυασμένες κοινέ μεταξύ των, των χωρών ε, και οτιδήποτε αφορά ε, την ιδιαιτησία γενικότερα αυτό είναι κύλι διαιτητικά δικαστήρια. Τα έχουμε συζητήσει πολύ τον τελευταίο καιρό, άρα θα πρέπει να βρεθεί κάποια άλλη λύση. Η άλλη λύση είναι αυτή που Πιστεύουμε ότι ένα τέτοιο, ένας τέτοιος μηχανισμός επίλυσης διαφορών ε, θα ε, ηρεμήσει κατά κάποιο τρόπο. Η κεντρική γραμμή, αν θέλετε, αυτής της δρομοδότησής μου είναι ότι θα πρέπει να βρεθεί ε, μια σωστή ισορροπία. Ανά σας πω και σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Δεν ξέρω αν κάποιο μέλο, αν κάποιος βουλευτής θέλει να πάρει το λόγο. Όχι από ό,τι φαίνεται νομοποίηση και λογοδοσία. ευαίσθητο. Πρόεδρος, να σας πληροφορήσω λοιπόν ότι μπορείτε να υποβάλλετε τροπολογίες μέχρι τις 29 Ιουνίου το μεσημέρι. Πάρα πολύ ωραία. Ολοκληρώσαμε λοιπόν ε, και την ε, μελέτη του σημείου 23. Το 24 έχει διαγραφεί. Ε, φτάνουμε στις 25, συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου. Έχουμε εδώ και τον ε, κύριο Φως και την κυρία Γκέπχαρτ, είναι οι δύο συν εισηγητές. Δεν ξέρω ποιος θέλει να πάρει πρώτο το λόγο. Κύριε Φως. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκεί τίθεται ακόμα θέμα διατυπώσεων, χρειάζεται κάποια προσπάθεια, αλλά μάλλον μπορώ να πω ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση τέρηση ή σε κάποιο μπροκάρισμα. Αφενός το θέμα των αγαθών ή τα προϊόντα embedded software να μπουν στην οδηγία για τις επιγραμμικές πωλήσει, ενώ εμείς ακόμη δεν μπορούμε την ε, οδηγία, είχαμε πει νομίζω μέχρι τον Οκτώβριο, ώστε μέχρι τον Οκτώβριο να έχουν γίνει τέτοια βήματα πρόοδου ώστε εν τέλει να μπορούμε να πούμε κάτι στην οδηγία μας εμείς το οποίο ωστόσο να μην συμβαδίζει ό,τι αφορά τις νομικές ε, συνέπειες με τις ρυθμίσεις για τα άλλα. Πρέπει να κινητοποιήσουμε το Συμβούλιο Υπουργών να προχωρήσει και με την ε, οδηγία επιγραμμικών πωλήσεων online sales ώστε να μπορέσουν εν τέλει και να προκύψουν από την εργασία του κάποια αποτελέσματα. Διότι το ιδεώδε θα ήταν και τα δύο πακέτα και οι δύο δέσμες ε, προ την λήξη της κοινοβουλευτική περίοδου. Και γι' αυτό ζητήσαμε από το Συμβούλιο ή δυνατόν μέχρι τον Οκτώβριο να καταλήξει